έναν πρόεδρο συνελεύσεως ε, να φέρεται με τέτοιο κομματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Γκόλνης. Θα μεταφέρω το μήνυμά σας στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Θα σας παρακαλούσα αγαπητοί συνάδελφοι να επανέλθει η τάξη στο Κοινοβούλιο, στην αίθουσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε τις ε, επεξηγήσεις ψήφου. Έχουμε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, πολλά αιτήματα. Παρακαλώ, ησυχάστε συνάδελφοι, γιατί πρέπει να το ακούσετε αυτό που λέω. Μπορούμε να ε, ε, συζητούμε μέχρι τις 14.45. Μετά θα πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουμε έτσι ώστε να προετοιμαστεί η αίθουσα για την ε, συνεδρίαση που ξεκινάει στις 3. Όσοι δεν μπορέσουν να πάρουν το λόγο θα στείλουν τις επεξηγήσεις τους γραπτά. Έκθεση Φερνάντες, δίνω το λόγο στην κυρία Ρουέδα. Ευχαριστώ πολύ. Τα θέματα τα οποία ε, αναφέρονται εδώ είναι αρκετά σημαντικά. Ωστόσο, εγώ ε, αποφάσισα να απόσχω σε αυτήν την ψηφοφορία, γιατί πιστεύω ε, ότι από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να βγει από το παρόν πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Χρειαζόμαστε ένα πραγματικά δυνατό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων επενδύσεων έτσι ώστε να μπορέσει να μειωθεί ε, το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων ε, και έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε οικονομική και κοινωνική συνοχή. Ε, υπάρχουν πολλά κενά γύρω από το πρόγραμμα Juncker. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε τις δημόσιες επενδύσεις και να σταματήσουμε ιδιωτικοποιήσεις που θα αφορούν δημόσια αγαθά όπως το νερό ή το ηλεκτρικό. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον κύριο Σμιτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ε, καταψηφίσαμε την έκθεση Φερνάντες και αν ρωτούσατε και τους Ευρωπαίους νομίζω πως θα απαντούσαν και εκείνοι όχι. Γιατί, όχι γιατί είμαστε κατά όλων αυτών των σωστών πραγμάτων που περιέχονται, επιχειρηματικότητα κτλ. Αλλά η μόνη απάντηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεγαλύτερος προϋπολογισμός και ήδη πόροι, παρά το ότι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κανένα ε, θεσμικό όργανο δεν έχει λιγότερη νομοποίηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πώς τολμάτε να τα λέτε αυτά στους ευρωπαίους πολίτες ότι θέλετε και άλλα λεφτά για μας. Και αυτό είναι το σκεπτικό αυτής της ε, έκθεσης. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Γι' αυτό και το καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ κύριος Πόλτσακ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, ψήφι, εγώ υποστήριξα αυτή την ε, έκθεση. Ήταν νομίζω πάρα πολύ σωστή αυτή η ψηφοφορία. Η έκθεση περιγράφει σωστά την κατάσταση στον τομέα του προπολογισμού. Θα ήθελα όμως να τονίσω δύο πράγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά. Το ένα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει πραγματικά να αναφερθούν γιατί πάνω το, είναι πάνω από το 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και επλήγησαν από την ε, κρίση. Και ο ρόλος των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να συνδυθεί με το διαρθρωτικό με τα διαρθρωτικά ταμεία που αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό μοχλό επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτές τις εκθέσεις και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτά τα οποία κάναμε. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Περνάμε τώρα στην καταπολέμηση της απάτης έκθεση 2013 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας. Ο κύριος Πως Πίσελ είναι ο πρώτος. Για ένα λεπτό. Όχι. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υποστήριξα αυτή την έκθεση διότι θεωρώ την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σημαντικό θέμα. Σημειώθηκε και σημαντική πρόοδος κατά τα άλλα. Και την, ε, τα επιβλαβή, τις πράξεις ε, όσον αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αυτές οι πράξεις διώχονται βάσει ποινικού κώδικα. Και έτσι λοιπόν και με τα κράτη-μέλη και με την ΕΕ προσάγονται οι υποθέσεις στα δικαστήρια. Είναι και καλή η περιγραφή των δραστηριοτήτων της Όλαφ. Ελπίζουμε ότι η Όλαφ όλο περισσότερο θα έχει τη δυνατότητα χρήσης ε, των δυνατοτήτων της για την προστασία των ε, οικονομικών συμφερών. Πρέπει να διαχέονται οι πληροφορίες ε, και αν υπάρχει αξιόπινη πράξη τότε θα, θα πρέπει σαφείς αποφάσεις δικαστικές να υλοποιούνται. Υποστηρίζουμε την έκθεση αυτή λοιπόν. Ευχαριστώ. Επόμενος Τζουφρέντα, παρακαλώ, κυρία Τζουφρέντα, ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα στοιχεία τα οποία είδαμε ε, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχει αυξηθεί κατά 14% το ποσοστό απάτη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Κύριο θύμα βεβαίως ε, αυτών των απατών είναι η πολιτική συνοχή. Ε, δηλαδή πρόκειται για χρήματα, για πόρους που αφαιρούνται από τα προγράμματα τα οποία θα συνέβαλαν στην ευημερία των πολιτών μας. Πολλές κινήσεις και πολλά προγράμματα ε, είναι, ε, ε, οφείλονται στην ελληπή γνώση των διαδικασιών και στην περιπλοκότητα αυτών των διαδικασιών. Ζητώ, ζητώ βεβαίως να καταπολεμηθούν με μεγάλη σοβαρότητα και με μεγάλη, και με μεγάλη αυστηρότητα όλες αυτές οι απάντησεις ε, οι οποίες ε, γίνονται από πρόθεση. Με την ίδια, με την ίδια όμως αυστηρότητα να κινηθούμε υπέρ αυτών που παραβίασαν χωρίς να το γνωρίζουν. Ε, επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Άντερσον, αλλά νομίζω ότι δεν είναι εδώ, οπότε ο κύριος Χέις για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα αυτή την ετήσια έκθεση γιατί αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των συνθήκων. Η Κομισιόν έχει ζητήσει κάθε χρόνο να υπάρχει μια ετήσια έκθεση η οποία να δείχνει ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα προφανή παραδείγματα απάτης όχι μονάχα στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο είναι βεβαίως τα λαθρέα προϊόντα καπνού 10 δις ευρώ ε, απώλεια εισοδήματος έχουμε κάθε χρόνο και επομένως ε, θα πρέπει να το δούμε αυτό από ε, πολύ ε, κοντά. 628 ε, εκατομμύρια ε, ε, κουτιά τσιγάρων έχουν διακινηθεί μόνο στην Ιρλανδία και πέρα από τις κατασχέσεις οι οποίες μπορεί να γίνονται στη δικιά μου χώρα ή και αλλού χρειάζεται μια πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στις δημόσιες αρχές, την αστυνομία, τα τελωνία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ευχαριστώ πολύ. Τίτσο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποκαλεί έκθεση όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων σε ΕΕ. Κύριο στόχο είναι να σταματήσουν οι παράνομε δραστηριότητε και να ενθαρρυνθεί η χρηστή διαχείριση. Σε αυτή την έκθεση για το 2013 τονίζεται ότι αρνητικέ επιπτώσει μειώθηκαν οι επιβλαβεί πράξει κατά 17%. Ταυτόχρονα όμω οι παραβάσει και παραβιάσει ε, ω περιπτώσει αυξάνονται μπορούμε να δούμε ότι το σύστημα λειτουργεί πλέον καλύτερα όσον αφορά την ανείχνευση παραβιάσεων και παραβάσεων. Όμως είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά για την πρόληψη. Θέλω να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτρέψω να εργαστούν εντονότερα ώστε να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα με την υπεύθυνη δράση και στάση και θα πρέπει τα πάντα να γίνουν όσον αφορά τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρχει φοροδιαφυγή και φοροαπάτη και ότι θα μειωθούν οι περιπτώσεις αυτές στο μέλλον. Ο επόμενος ομιλητής, ομιλητής κύριος Τζάρξ δεν παρίσταται. Μέσερ Σμιτ παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ και είναι ασυνήθιστο για μένα ωστόσο όμως ε, να ενθαρρύνω τους πολίτες ε, να αναγνώσουν αυτές, αυτή την έκθεση των ε, θεσμικών οργάνων μια έκθεση όμως που θα έπρεπε να αναγνωστεί είναι η έκθεση του Ελεκτικού Συμβουλίου και μπορούν οι άνθρωποι να δουν, οι πολίτες να δουν το τι γίνεται και είναι εκπληκτικό πόσο μικρός βαθμός ελέγχου υπάρχει Εκείνο το οποίο εκπλήσει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αλλάζει τις πολιτικές της ε, και δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μια πειθαρχημένη προσέγγιση ώστε να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια των φορολογουμένων με πιο πειθαρχημένο και συντονισμένο τρόπο, όπως απαιτείται σε σχέση με τα κράτη-μέλη για παράδειγμα. Υπάρχουν λοιπόν ολόκληρα ταξίδια και προσπάθειες που γίνονται για να, να προσαυξηθεί η ε, προσέγγιση των πολιτών στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Ασυνήθιστο είναι να συμβαίνουν αυτές οι περιπτώσεις παράβασης των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόλτσακ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης ε, που την υπερψήφισα το θέμα των απατών θα ήθελα να τονίσουμε, να τονιστεί ιδιαίτερα και να δούμε τι γίνεται με τις πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αληθεύει ότι όσον αφορά τα ποσά συνολικά έχουν μειωθεί οι απάτες, όμως οι περιπτώσεις ε, σε συχνότητα απατών αυξάνονται οι περιπτώσεις αυτές. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω και κάτι για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και στο επίπεδο κιόλας ε, της ε, ε, συγχρηματοδότησης με εθνικά κονδύλια. Στα περιφερειακά για παράδειγμα προγράμματα το βλέπουμε αυτό. Υπάρχει η περίπτωση αυτή κατάχρησης κονδυλίων και συμβαίνει να μην υπάρχουν πολλές φορές έλεγχοι και σε σχέση με την τσεχική δημοκρατία ολόκληρη, όλη η μέθοδος μεθοδολογικά έπρεπε να τροποποιηθεί. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν θα πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα και για να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τα εθνικά προγράμματα που θα τα αντικαταστήσουν. Um, Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου για την έκθεση πρόοδου για το Μαυροβούνιο. Παρακαλώ καπούτο ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Μαυροβούνιο έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλε πρόοδους όσον αφορά την ένταξη, την πορεία εντάξεως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ήδη ανοίξει 16 κεφάλαια διαπραγμάτευσης, ε, μεταξύ των οποίων και μερικά πολύ σημαντικά. επίση, με πολύ ενεργητικό τρόπο ε, και πολύ θετικό τρόπο έχει, ξεκινήσει η διαδικασία αυτή με το Μαυροβούνιο. Και αυτή τη στιγμή φέρεται πάρα πολύ καλά όσον αφορά την διεθνή αντιμετώπιση της απειλής της τρομοκρατίας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σωστό να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις και γι' αυτό ακριβώς υπερψήφιση. Thank you. Our next speaker... Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπόγκοβιτς, για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο ξεκίνησαν το 2012 και μέχρι στιγμής έχουμε ολοκληρώσει τα 16 από τα 32 κεφάλαια, δύο έχουν πλήσει προσωρινά, οπότε το Μαυροβούνιο βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας, της ανάπτυξης. Βλέπουμε ήδη αποτελέσματα στο Μαυροβούνιο. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν όπως και στις άλλες υποψήφιες ε, χώρες. Ε, εξάλλου παρόμοια είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο. Υπάρχουν κάποια ζητήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, όλα αυτά είναι τομείς ε, που είναι προβληματικοί για ολόκληρη την περιοχή. Εγώ λοιπόν θα ήθελα μια καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους του Μαυροβουνίου, αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να γίνει κάτι και με την γενικότερη κοινωνική οργάνωση. Ευχαριστώ κύριο Τζαμπάσκι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ στήριξα την έκθεση αυτή γιατί είναι αντικειμενική και δείχνει την πρόοδρο του Μαυροβουνίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω. οι αδυναμίες του Μαυροβουνίου επίσης φαίνονται εδώ, σχετίζονται με την ελευθερία των ΜΜΕ, της έκφρασης, υπάρχουν κάποια πράγματα που αφορούν τις σχέσεις με την Ουκρανία, αλλά συνολικά το Μαυροβούνιο είναι πρώτο πόρος όταν μιλάμε για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Στο Μαυροβούνιο υπάρχει πλήρης ε, ομοφωνία όταν μιλάμε για την κρίση στην Ουκρανία ή την αντιτρομοκρατική νομοθεσία που αφορά το Ισλαμικό κράτος στο Μαυροβούνιο είναι σαφής η στάση τους απέναντι σε όσους δραστηριοποιούνται στο πλευρό του Ισλαμικού κράτους. Γι' αυτό ακριβώς προστήριξα αυτή την έκθεση γιατί είναι αντικειμενική. Ευχαριστώ. Η κυρία Πετήρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ υποψήφισα αυτό το ψήφισμα για το 2014 και το Μαυροβούνιο γιατί σε πάρα πολλά σημεία λέει ξεκάθαρα πως έχει γίνει πρόοδος αλλά επισημαίνει και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο. Θα ήθελα επίσης να τονίσω όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τα διαπραγματευτικά κεφάλαια 23 και 24 και αφορούν κυρίως το κράτος δικαίου, την αποτελεσματική δικαιοσύνη, καταπολέμηση της διαφθοράς, ελευθερία του τύπου, καθώς και κανονισμούς για την ε, χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, καθώς επίσης ε, και τις ε, αποζημιώσεις στα θύματα του πολέμου και την Κροατία. Επίσης, μιλάει για την δημιουργία μιας ατμόσφαιρας ανοχής όσον αφορά τις ε, μειονότητες. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν οι αρχές αυτές να προστατεύσουν τον πολυεθνικό χαρακτήρα της Μπόκα Κότευσκα και να συνεργαστούν στενά με τις γειτονικές χώρες. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση 2014 για την Πουγουδουμού. Δίνω τον λόγο στην κυρία Μπόρζαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Στήριξα την έκθεση αυτή γιατί υπάρχουν δύο σημαντικά πολιτικά μηνύματα. Πρώτον, ότι η Μακεδονία ήταν η πρώτη η οποία ε, ε, σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις, υπορεώθηκε μάλλον λόγω ενός διμερούς θέματος με την ε, Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά η ίδια η Κομισιόν προτείνει την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων ούτως ή ένα δεύτερο ζήτημα είναι το θέμα της ε, δημόσιας διακυβέρνησης στη Μακεδονία. Ε, μονάχα λίγες ε, είναι οι κατηγορίες οι οποίες αφορούν φόβο για παρανομίες στον πολιτικό βίο της χώρας. Αλλά βεβαίως έστω και αν ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτών των κατηγοριών ε, να ισχύει, τότε οπωσδήποτε το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λοιπόν θα ζητώ από τις αρχές να το κοιτάξουν. Ευχαριστώ πολύ. Πόγκοβιτς για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Το ψήφισμα αυτό σε σχέση με την Μακεδονία που υποστηρίζουμε διότι ταυτοποιείται η κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου ρόζινη, ρόδινη και η Μακεδονία θα έπρεπε να κάνει βήματα προς την ορθή κατεύθυνση τα προβλήματα θα έπρεπε το δυνατόν ταχύτερο να επιληθούν, ώστε οι διαπραγματεύσεις να μπορέσουν να ξεκινήσουν επιτέλους. Η σημερινή πολιτική κατάσταση στην Μακεδονία είναι προβληματική και αν καθυστερήσουν οι διαπραγματεύσεις μπορεί να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη έκδηλη κρίση στην χώρα αυτή. Θα έπρεπε να υποστηρίξουμε την επιθυμία να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε η κατάσταση να επιδεινωθεί περαιτέρω και να αποσταθεροποιηθεί. Θα πρέπει <clears throat> σε σχέση με ένα διάλογο να ξεκινήσει για τη σταθεροποίηση της περιοχής. Ο κύριος Τζαμπάσκι παρακαλώ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, υποστήριξα αυτή την έκθεση είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο αποστέλλεται στην κυβέρνηση των Σκοπίων. Πρέπει να επιληθούν διμερεί προβλήματα. Η σύμβαση, συνθήκη σε σχέση με την Βουλγαρία θα πρέπει να ε, προχωρήσει και να γίνει σεβαστή και θα πρέπει σε σχέση με τα μέσα του τύπου και τα δικαιώματα των πολιτών να είναι σεβαστά. Πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους οι πολίτες στη χώρα αυτή. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται σε ένα έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, με τον όρο πολίτες της Μακεδονίας ε, και αναφέρεται εδώ και το θέμα της Βουλγαρίας. Θα πρέπει να μπορέσει να υπάρξει δυνατότητα αυτής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ε, Πετήρ παρακαλώ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Υποστήριξα και μάλιστα με την αλληλεγγύη που εκφράζουμε εναντί της Μακεδονίας ε, προσκαλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξεύρουν μία λύση μετά από πολλές αποτυχίες ώστε να ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία ενώ η διμερής διαφορά πρέπει ταυτόχρονα σε παράλληλη τροχιά να επιληθεί περίμενε πάνω από 10 χρόνια η Μακεδονία λόγω του προβλήματος για την ονομασία της με την Ελλάδα και αυτό είναι πολύ αποθαρρυντικό και απογοητευτικό για τους πολίτες της. Η Κροατία δίνει ένα υπόδειγμα, ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να εφαρμοστεί και στη Μακεδονία. Και πάλι προσκαλώ το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν αυτά τα θετικά παραδείγματα από τον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων και κατεπηγόντως να εξευρεθεί δυνατότητα να αρχίσει αρχίσουν επίσημα οι διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία και την ΕΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στην έκθεση πρόοδου για την Σερβία. Ο κύριος Ποσπίσουλ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε ως ε, μέλος της Επιτροπής ε, για την Σερβία χαιρετίζω την έκθεση αυτή που περιγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πάρα πολλά μέτωπα. Είναι μια έκθεση ισορροπημένη γιατί αναφέρονται και τα προβλήματα που απασχολούν ακόμα την Σερβία. Εγώ ασχολούμαι κυρίως με τη δικαιοσύνη και με ενδιαφέρουν τα ζητήματα αυτά δικαιοσύνης, αστυνομίας, διαφθοράς. Παρόλες τις ε, προσπάθειες ε, πρέπει να γίνουν ακόμα βελτιώσεις για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα κράτος ε, δικαίου. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι σαφές ότι υπάρχει αυτή η έκκληση εντός της έκθεσης. Χωρίς κράτος δικαίου δεν είναι δυνατόν να γίνει κράτος μέλος ε, η Σερβία. Θα πρέπει λοιπόν η μεταρρύθμιση αυτή να γίνει και είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ δύσκολη και όλες οι πρώην κομμουνιστικές χώρες ε, θα έπρεπε να μπορούν να την εφαρμόσουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το ψήφισμα για την πρόοδο της Σερβίας ε, το υποστήριξα με ιδιαίτερη χαρά. Γίνεται λόγος για προσπάθειες της σερβικής κυβέρνησης ε, για αυτό το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και για, για καλύτερες ε, σχέσεις με κράτη της περιοχής αυτής του κόσμου και για πρόοδο όσον αφορά το κράτος δικαίου που θα αποβαίνει υπέρ της Ευρώπη. έχω την πεποίθηση ότι το αξίζουν οι πολίτες της Σερβίας να εκφραστεί η αλληλεγγύη της Ευρώπης προς αυτούς. Και έτσι λοιπόν να προετοιμαστεί η χώρα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι ικανή να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες της σερβικής κυβέρνησης και του πληθυσμού των πολιτών της Σερβίας για την ακολούθηση αυτής της πορείας πρέπει να υποστηριχθεί οπωσδήποτε αυτή η πρωτοβουλία με διαφορετικά μέσα και εργαλεία για την υποστήριξη και χρηματοοικονομική υποστήριξη ώστε να βοηθηθεί η Σερβία καθοδόν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ευχαριστώ κύριο Τζαμπάσκι. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Υποστήριξα και εγώ αυτή την έκθεση. Όμως υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την κυβέρνηση. Τον σεβασμό των κανόνων του παιχνιδιού και των κανόνων των μειονοτήτων, τον σεβασμό των μειονοτήτων. Κάθε μειονότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να ε, διδάσκεται και να διδάσκεται διδάσκει την γλώσσα της. Ε, ιδιαίτερα για την βουλγαρική μειονότητα ε, που αναγνωρίζεται από την ίδια τη Σερβία και που υπάρχουν πολλοί φραγμοί και εμπόδια για αυτή την μειονότητα. Πρέπει ένα πολύ σαφές μήνυμα λοιπόν να αποσταλεί με αυτόν τον τρόπο έτσι στη Σερβία και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Πέτια παρακαλώ. Εγώ στήριξα στήριξα την έκθεση αυτή όσον αφορά την έκθεση προόδρου ε, της Σερβίας του κ. Μακάλιστερ γιατί πιστεύω ότι μεταφέρει αυτό το ε, κύριο μήνυμα ότι θα πρέπει να προχωρήσει η Σερβία ε, στην διαδικασία ενσωμάτωσής της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Σερβία έτσι ώστε να λάβει υπόψη διάφορες προβληματικές Κυρίω ε, Κυρίως εδώ αναφέρομαι στους αγνοούμενους ε, και στους Κροάτες της Βοηβοντίνας. Ε, νομίζω λοιπόν ότι τώρα διαπιστώνουμε πλέον πόσο προβληματική είναι η κατάσταση στην Σερβία η οποία παραβιάζει την αρχή της καθολικής δικαιοσύνης καθώς επίσης και τις αρχές οι οποίες από αυτήν απορρέουν. Η Σερβία δεν θέλει να τα καταλάβει όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά θα ήθελα να τους ε, καλέσω να ε, ε, απαλείψουν τα άρθρα 2 και 3 και βεβαίως να δίνουν την δυνατότητα σε όλους να έχουν την ίδια δικαιοσύνη. Ζητώ συγγνώμη δεν σας είχα δει συνάδελφε. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην οικονομική και πολιτική ζωή είναι αυτονόητο ότι η Σερβία ανήκει άρρηκτα στην Ευρώπη. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο ο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις προσπάθειες ε, να προσεγγίσει και να ενταχθεί η Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να γνωρίζει η Σερβία ότι τότε μόνο θα καταστεί αυτό εφικτό όταν θα έχει υπάρξει συμφιλίωση προηγούμενα με όλες τις εθνικές και εθνοτικέ μειονότητες. Ε, λαός που έχει υποφέρει τόσο πολύ θα πρέπει πραγματικά με αυτόν τον τρόπο να ακολουθεί την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω αυτή την έκθεση και ελπίζω ότι θα υπάρξουν περαιτέρω πρόοδοι. Ε, δεν είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι υποχρεωτικές αυτές οι ε, αλλαγές. Δεν είναι υποχρεωτικό με πίεση εκ των έξω να επιτευχθούν αυτές οι πρόοδοι. Είναι αναγκαίο εκ των έσω να επιτευχθούν και να αποτελέσει ένα ε, παράδειγμα για άλλες ε, χώρες. Διότι βλέπουμε στην Ρουμανία και αλλού υπήρξαν οπισθοδρομήσεις. σόλτες παρακαλώ στη συνέχεια. Πρέπει να ομολογήσω και να πω ότι κατά την παρακολούθηση της Σερβίας καθώς η Σερβία προσεγγίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα τελευταία έτη έκανε σημαντικές πρόοδους σε, διαφορετικούς, σε διάφορους τομείς η Σερβία μεταρρυθμίσεις επετέφθησαν για παράδειγμα στον τομέα της δικαιοσύνης μεταρρυθμίσεις που είναι πολύ σημαντικές για να μπορέσει να ενταχθεί η Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αληθεύει όμως επίσης ότι κάποιοι εξωτερικοί λόγοι και ε, γεγονότα δεν ήταν ιδιαίτερα θετικά για παράδειγμα οι πλημμύρες ε, που έπληξαν την ε, Σερβία και την ευρύτερη περιοχή της η Σερβία διανύει μια περίοδο δυσχερέστατη από οικονομικής πλευράς πρέπει να υπάρχει υπάρξει δράση άμεσα ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξει αυτή η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τη Σερβία. Και πρέπει να δούμε και τον ρόλο των ομόρων κρατών. Και όταν κάνουμε λόγο για τη Σερβία, πρέπει να επιδειχθεί αλληλεγγύη και πρέπει να υπάρξει βοήθεια που θα δοθεί. Σα ευχαριστώ, συνάδελφοι. Περνάμε τώρα στι αιτιολογήσει ψήφου για το Κωσίφο Πέδιο. Προτού γίνει αυτό, θα ήθελα να κάνω μια ε, αναγγελία να πω ότι έπρεπε να ολοκληρώσουμε παρατέτατο. Και τώρα θα πάρουμε μόνο αιτιολογήσεις ψήφου για το κοσυφοπέδιο και την έκθεση Ντάριους Ροζάτη, ώστε να μπορέσει να τηρηθεί το χρονικό όριο. Σας διασφαλίζουμε ότι θα δοθεί η δυνατότητα να κάνετε τις αιτιολογήσεις ψήφου αύριο, όταν θα αρχίσει η περίοδος, ε, η ώρα των επεξηγήσεων. Περνάμε στην, ε, στο κοσυφοπέδιο. Έχει τον λόγο ο κύριος Μπόγκοβιτς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ το ψήφισμα για την διαδικασία της ολοκλήρωσης του Κωσυφοπεδίου το στήριξα γιατί μας δίνει μια γενική εικόνα του τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρει βεβαίως και τα προβλήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το κοσυφοπέδιο. Βλέπουμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, πως ε, οι άνθρωποι πλέον βλέπουν πως το μέλλον, το μέλλον τους θα είναι δύσκολο στην ε, χώρα τους γιατί υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα που δεν λειτουργούν. Το πρόβλημα όμως αυτό της εξόδου είναι ε, οπωσδήποτε ανησυχητικό αλλά και ενδεικτικό της ε, ανησυχητικής ε, κατάστασης και βεβαίως προβληματίζει και τις γειτονικέ και άλλες χώρες. Μιλάμε κυρίως για εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται την ε, κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στήριξα αυτή την έκθεση γιατί η εισηγήτρια, η κυρία Λούνατσεκ ε, συνέταξε μια ισορροπημένη έκθεση. Βεβαίως υπάρχουν πολλά προβλήματα στο κοσφοπέδιο που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα, το εμπόριο ναρκωτικών, οικονομικά προβλήματα που αναγκάζουν τον κόσμο να φύγει. Και εδώ πέρα βεβαίως εμείς ζητάμε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Αυτός είναι σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει το κοσμοπέδιο αν θέλει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Οπότε κάτι κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό στήριξα αυτή την έκθεση. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι αποδεκτό το κείμενο αυτό, διότι απλά δεν λαμβάνει υπόψη ε, τα, τα προβλήματα των Σέρβων τόσο προσφυλών στον Βίκτορα Ουγκό. Ε, η Σερβία είναι μια το Κωσυφοπέδιο υποτίθεται θα ήταν μια χώρα ε, η οποία υποτίθεται, στην οποία υποτίθεται ότι συμβιώνουν αρμονικά Σέρβοι, Αλβανοί κλπ. Αλλά παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ακριβώς το αντίθετο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας τίποτα δεν έχει καταλάβει σωστά από την κατάσταση σε αυτήν την ε, περιοχή. Η Ουτσεκά έχει προχωρήσει σαν τρομοκρατική οργάνωση και ακόμα και το γεγονός ότι Ορισμένοι θεωρούν ότι το κοσυφοπαίδιο θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι ε, οι ίδιοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τον απόλυτο εντετερμινισμό αυτή τη περίπλοκη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστήριξε αυτό το ψήφισμα για το κοσυφοπαίδιο, διότι η βούληση που εκφράζεται ελεύθερα, από τους πολίτες και μάλιστα με ολοκλήρωση και με ελευθερία, με ειρήνη και σταθερότητα είναι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστορία ε, ε, του Κωσυφοπεδίου, τις ιδέες ε, της εδαφικής επικράτειας και της ελευθερίας συνεχίζουν χωρίς να γίνεται αντιληπτό ότι χρειαζόμαστε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη. Ευρώπη ενωμένη για να είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις με ελεύθερη ε, συνεργασία των επιμέρους μερών, των πολιτών. Ένα χώρο για τόσο ευαίσθητα θέματα όπως ε, για την εθνική ταυτότητα θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν ε, η περιφερειακή εδαφικότητα να μπορέσει να ληφθεί υπόψη. Μια άλλη αρχή που πρέπει να επανεξεταστεί. Ευχαριστώ. Περνάμε στις τελικές επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Ροζάτη. Για ένα λεπτό Τζουφρέντα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση γιατί όλοι πρέπει ε, να καταλάβουμε και να το δεχτούμε ότι η ανάκαμψη που περιμέναμε δυστυχώς δεν πρόκειται να έρθει. Οι τρεις προτεραιότητες ε, μας βρίσκουν ε, σύμφωνους και οπωσδήποτε θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη. Είναι σημαντικό πάντως να υπογραμμίσουμε ότι στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να λείπει η ευελιξία. Οι παρεμβάσεις στους προϋπολογισμούς δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους προϋπολογισμούς και σίγουρα να μην αποτελούν αντικίνητρο για τις επενδύσεις. Οι μικρές εταιρείες οπωσδήποτε έχουν ακόμα πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία όσον αφορά την πρόσβαση στην πίστη και την χρηματοδότηση. Ε, υπάρχουν χώρες ε, οι οποίες ακόμα αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, πολύ μακριά από την τυποποίηση βρίσκονται. Επίσης, ε, το να περιμένουμε απλώς να πέσει από τον ουρανό η ανάπτυξη είναι κάτι αφελές, αλλά ε, θα πρέπει να ξέρουμε τι θα διορθώσουμε έτσι ώστε να προχωρήσουμε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ στήριξα την έκθεση αυτή γιατί καλωσορίζω τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η οποία ε, υποστηρίζει, βασίζεται κυρίως στην ε, ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει οι επενδύσεις να είναι ισορροπημένες και φιλικές προς την ανάπτυξη. Ωστόσο πιστεύω ότι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τα ίδια τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Επίσης να λάβει υπόψη και τις χώρες οι οποίες έχουν μειώσει το υπερβολικό ε, έλλειμμα. Η κυρία Μάλετη, της ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, οι τρεις πυλώνες στις οποίους βασίζεται η ανάπτυξη είναι μεταρρυθμίσεις, εξυγένση των δημοσίων οικονομικών και επενδύσεις. Επενδύσεις, έρευνα και ανάπτυξη, σε εκπαίδευση, σε εξυγχρονισμό, φθηνότερη ενέργεια, όλα αυτά είναι σημαντικά για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Οι επενδύσεις λείπουν γιατί δεν ε, υπάρχει διάθεση να αναλάβει κανείς ε, κινδύνους και οι χρηματαγορές μας είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένες. Μπορεί λοιπόν το κενό αυτό να κλείσει αν ανοίξουμε νέες δυνατότητες να δοθούν δάνεια σε επιχειρηματίες. Η έκθεση αυτή δείχνει πως οι θετικοί και γενναίοι κυβερνήτες μπορεί να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον τους. Γι' αυτό και εγώ είμαι αισιόδοξος. Αισιόδοξη, με συγχωρείτε. Η κυρία Κινίτση. Ευχαριστώ πολύ Πολλές και μεγάλες οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που οπωσδήποτε επιβραδύνουν ε, την ε, όθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν προβλέπεται μια σχετική ανάκαμψη ε, για το 2015 και το 2016. Προώθηση όμως και πρόδρος η οποία αναφέρεται σε στοιχεία τα οποία ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει πραγματικά την πορεία τους. Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι προϋπολογισμοί έτσι ώστε να, γίνει, να δοθεί δυνατότητα στην ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υπάρχει σωστό σχεδιασμός των, ε, ε, των επενδύσεων έτσι ώστε ε, ταυτοχρόνως να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας ή, και να, ταυτόχρονα να βελτιωθούν οι δυνατότητες εργασίας κυρίως αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της νεανικής ανεργίας και των μακροχρονίων άνεργων. Θεωρώ ότι η έκθεση προς την κατεύθυνση πηγαίνει και γι' αυτό την υπερβολή. Ευχαριστώ ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την έκθεση αυτή. Και αυτό όχι γιατί δεν συμφωνώ με τους αριθμούς. Βεβαίως μπορεί κανείς να ε, συζητήσει και τους αριθμούς και το περιεχόμενο. Απλώς θεωρώ ότι ε, στην έκθεση διαφαινόμενες προοπτικές είναι παντελώς ε, λανθασμένες. Η ανάπτυξη στον κόσμο ολόκληρο είναι πιο σημαντική στην ε, ε, Ευρώπη ε, και στην Ευρώπη περισσότερο από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από ότι στην Ευρωζώνη. Επομένως νομίζω ότι το πρόβλημα είναι το ευρώ και θα πρέπει κάποτε να το κατανοήσουμε έτσι ώστε να κλείσουμε αυτό το ευρώ έξω από την πόρτα μας. Ε, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λένε μερικοί, καταλαβαίνω την άποψή τους αλλά νομίζω ότι το ευρώ ήταν ένα κακό πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να ρίξουμε στο σκουπίδο Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάλτσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, εγώ το απορρίπτω και επί της ε, αρχής, αλλά και για λόγους ε, θεωρητικούς. Θα πρέπει πραγματικά η κάθε κυβέρνηση να μπορεί να λειτουργεί ως ε, τέτοια. Γι' αυτό βλέπουμε πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία καμουφλάρονται και μιλάμε για στενότερη οικονομική συνεργασία και στην ουσία επαγορεύουμε στα κράτη τι πρέπει να κάνουν και τι να βάλουν στον προϋπολογισμό τους. Και μετά, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, γίνονται συζητήσεις και ε, μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν τα αποδέχεται αυτά ή όχι. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πως το μέτρο αυτό λέει στα κράτη τι μπορούν να κάνουν. Έτσι παραβιάζεται η, τα κυριαρχικά δικαιώματα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Οι υπόλοιπε επεξηγήσεις ψήφου αύριο μετά την ψηφοφορία διακόπτουμε μέχρι τις 3.